Η κυρία Πρόεδρος. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επαναλαμβάνεται η συνεδρίαση. Τα συνοπτικά πρακτικά της θεσινής συνεδρίασης και τα κείμενα που εγκρίθηκαν σας έχουν διανεμηθεί. Ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχουν παρατηρήσεις. Οπότε θεωρώ ότι τα συνοπτικά πρακτικά εγκρίνονται. Το επόμενο σημείο στην ε, ημερήσια διάταξη είναι η κοινή συζήτηση σχετικά με τη μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής, σύμφωνα με το άρθρο 70α του κανονισμού.